Ε, Σύνοδο, Έχουμε τώρα στην ημερήσια διάταξη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής, είπα της εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας που θα μας μιλήσει για την κατάσταση στην Αίγυπτο. Θα σας ενημερώνω ότι εν ώψη της ε, καθυστέρησης που έχουμε δεν θα γίνει κατσδιά και δεν θα δεχτώ γαλάζιες κάρτες. Κυρία Μογκερίνη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε για την κατάσταση στην Αίγυπτο ουσιαστικά είναι μια χρονική περίοδος που είναι συμβολική σημασίας. Αν δούμε τι έγινε πριν τέσσερα χρόνια, βρισκόταν ε, ακριβώς ε, μπροστά σε μια επανάσταση η Αίγυπτος. Κατέβαιναν στους δρόμους διαδηλώνοντας για την αξιοπρέπεια και τη δικαιοσύνη οι πολίτες και για τα νόμιμα πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματά τους. Βοήθησε η Ευρωπαϊκή Ένωση την Αίγυπτο και τον λαό της υποστηρίζοντας τα αιτήματα αυτά με δράσεις. Τέσσερα χρόνια μετά, σήμερα, βρίσκεται σε μια πολιτική μετάβαση η Αίγυπτος. Και μετά από την ε, αποπομπή του Προέδρου Μόση συνεχίζεται αυτή η μεταβατική περίοδος και θα είναι ένα κρίσιμο βήμα για την, ε, το συνταγματικό χάρτη της Αιγύπτου αυτή η περίοδος. Δύο βήματα έχουν επιτευχθεί ένα νέο σύνταγμα και η εκλογή ενό νέου Προέδρου. Και τα δύο βήματα αυτά παρακολουθήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση με μια αποστολή για τις προεδρικές εκλογές το Μάιο. Μια αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετείχε επίσης. Τώρα θα θέλαμε να δούμε την αποστο... τις συστάσεις της αποστολής ε, να υλοποιούνται, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ε, υποεξέλιξη εκλογές είναι, υπάρχουν ε, πολλές δυσκολίες και αποφασίσαμε να μην στείλουμε μια πλήρη αποστολή αυτή τη φορά, αλλά να χρησιμοποιηθεί μιας μικρότερης κλίμακας ε, όργανο και να αξιολογηθεί η εκλογική διαδικασία, ακόμα και το πολιτικό περιβάλλον και η εκστρατεία η προεκλογική. Ο πίνακας των συστάσεων θα δώσει την δυνατότητα να εμπλακούμε επικοδομητικά με τις αρχές για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και προσπάθειες για τις μεταρρυθμίσεις. Η δημοκρατία πάει πιο πέρα από τις εκλογές και το γνωρίζουμε πολύ καλά. Έχει ρόλο κλειδί το Κοινοβούλιο για να διαδραματίσει το ρόλο αυτό για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που αναμένονται και τη μεταρρύθμιση για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, και ένα νομικό πλαίσιο και την συμμετοχή όσον αφορά ένα νέο σύνταγμα οι κοινοβουλευτικέ εκλογέ είναι ένα σημαντικό βήμα για να υπάρξει μια ευρεία βάση της πολιτική εμπλοκή που θα διασφαλίζει θεμελιώδη δικαιώματα, ελευθερίε, ασφάλεια, οικονομικέ μεταρρυθμίσει για την κοινωνία. Ανοιχτή πολιτική εμπλοκή και συζητήσει που θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της ριζοσπαστικοποίησης. Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα της ασφάλειας και της κατάστασης της χερσονήσου του Σινά. Είπαμε πάντα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνδράμει την Αίγυπτο και θα την βοηθήσει στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Και σε σχέση με τον ειδικό απεσταλμένο για αυτά τα θέματα εξετάζουμε τον διάλογο για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και για την ασφάλεια και είναι προς το συμφέρον και της Αιγύπτου αλλά και προς το συμφέρον της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια και είναι πολύ ευάλωτη η κατάσταση εκεί, τουλάχιστον ευάλωτη. Καλωσορίζουμε και καλωσορίσαμε την ανάδυση της Αιγύπτου ως ενός σημαντικού περιφερειακού ε, παίκτη. Είναι σημαντικός ο ρόλος ε, της Αιγύπτου όσον αφορά την εκεχηρία στη Γάζα κατά το, την περίοδο του καλοκαιριού και πιο πρόσφατα σε σχέση με την σύνοδο για την Γάζα και την ανοικοδόμηση που έγινε στο Κάιρο πρόσφατα. Επιπλέον η Αίγυπτος είναι ένας σημαντικός παίκτη στην εξωτερική πολιτική και για την Αφρικανική Ένωση και για τον Αραβικό Σύνδεσμο, τα Αραβικά κράτη και για το θέμα των υδάτων του Νείλου και με την Αιθιοπία για τη ρύθμιση αυτού του θέματος και βρίσκεται ακόμα σε μια πολιτική μετάβαση και αντιμετωπίζει θέματα ασφάλειας η Αίγυπτος και χρειάζεται συνδρομή και βοήθεια για τα οικονομικά της θέματα και την ανάπτυξή της. Τα βήματα που έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση βαίνουν προς την ορθή κατεύθυνση. Σημαντικές ε, μεταρρυθμίσεις έχουν γίνει όσον αφορά τις επιδοτήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες της Αιγύπτου για κοινωνικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Θα συμμετάσχουμε και στην Διεθνή Σύνοδο χορηγών ε, που θα γίνει τον Μάρτιο. Επικεντρώνουμε την υποστήριξή μας στο κοινωνικό-οικονομικό τομέα για να βοηθήσουμε να βελτιωθεί η κατάσταση της Αιγύπτου για τους πιο ευάλωτους κατοίκους αυτής της χώρας. Αυτές οι προκλήσεις συνολικά και η μετάβαση η πολιτική δεν μπορούν να επιτρέψουν κανένα συμβιβασμό για τα δικαιώματα του ανθρώπου στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτος πρέπει να ρυθμίσει τα θέματα των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των δικαιωμάτων εκείνων που έχουν διαφορετική άποψη και είναι αντιφρονούντες. Πάρα πολλά από τα θέματα τα οποία προαναφέρατε εσείς στο δικό σας ψήφισμα για την ελευθερία της έκφρασης δεν έχουν ακόμα ρυθμιστεί και διευθετηθεί στην Αίγυπτο. Τον προηγούμενο Δεκέμβριο είδαμε μια νέα απόφαση δικαστηρίων το θέμα δηλαδή των ε, ε, καταδικών σε θάνατο ε, πολλών αδελφών μουσουλμάνων. Και θα πρέπει να τονίσουμε ότι πρέπει να διασφαλιστεί μια δίκαια δίκη και να διασφαλιστούν τα δικαιώματα αυτών των ατόμων. Το θέμα της δικαιοσύνης λοιπόν και της μεταρρύθμισης της είναι σημαντικό. Μια άλλη ανησυχία και που όπως ε, αναφέρουμε σε σχέση με την τοποθέτησή μας είναι η απουσία λογοδότησης όχι μόνο οι διώξει των αδερφών μουσουλμάνων αλλά και των πολιτικών αντιπάλων και των πολιτικών ακτιβιστών είναι θέματα που παίρνουν πολύ δυσανάλογες διαστάσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες που καταδικάζονται από στρατοδικία και βρίσκεται εδώ το εκτελεστικό έχει εξουσίες υπερβολικές και βλέπουμε ότι όλα αυτά δεν συνάδουν ε, με τις ε, ρήτρες που πρέπει να είναι σεβαστές. Πάντα θα αναφέρουμε αυτά τα θέματα ώστε να μπορέσουν να διευθετηθούν σε σχέση με τους Αιγύπτιους. Είναι σημαντικά τα θέματα των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του ειδικού απεσταλμένου Λαμπρινίδη που διαρκώς θίγει αυτό το θέμα με τις Αιγυπτιακές αρχές και κατά την ε, επίσκεψη που ε, ε, σχεδιάζεται στην, προβλέπεται στην Αίγυπτο. Δεν θα πρέπει λοιπόν εδώ να θεωρηθεί κάποια άλλη εναλλακτική λύση ότι θα ήταν εφικτή. Πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε με τον καλύτερο τρόπο την επίσκεψη επίτευξη αυτού του εγχειρήματος. Έχει όπως και όλοι οι ε, εταίροι μας ε, της, ε, στη Μεσογειακή εταιρική σχέση προς τον Νότο έχει πλήρη συνδρομή από εμάς η, Ευ, Αίγυπτος. Θα πρέπει να αναδιαπραγματευτούμε πολλά τέτοια θέματα ώστε να μπορέσει να ληφθεί υπόψη η πραγματικότητα επιτόπου. Θα παρακολουθήσουμε τις κοινοβουλευτικές εκλογές με τους επαΐοντές μας όπως ανέφερα. Θα παρακολουθήσουμε την περαιτέρω εφαρμογή του συντάγματος και των μεταρρυθμίσεων και δεδομένων των κοινοβουλευτικών εκλογών και την ελευθερία του τύπου και των μέσων. Και έτσι λοιπόν με τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να βοηθηθεί η Αίγυπτος και θα συνεργαστούμε με την Αίγυπτο. Επίσης ε, με δικές μας προσπάθειες από τη δική μας πλευρά για τα θέματα ασφάλειας που μας αφορούν εμάς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Αντιπρόεδρε. Ο κύριος Πρέντα. Σας ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κυρία Αντιπρόεδρε για τα όσα μας είπατε. Καταρχήν θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια σε σχέση με τη θέση της ομάδας του ΕΛΚ για αυτά τα θέματα και σε σχέση με το ψήφισμα που διαπραγματευθήκαμε μαζί με τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες. Έχουμε μακρύ και λεπτομερές κείμενο και αυτό γιατί θέλαμε να καλύψουμε όλα όσα συνέβησαν από τον ε, Ιούλιο του 2014 όταν υιοθετήσαμε το τελευταίο μας ψήφισμα για την Αίγυπτο. Αυτό σήμαινε ότι δεν ήταν 100% ακριβή τα στοιχεία που είχαμε. Όμως το κείμενο αυτό θα πρέπει να το δούμε στο σωστό πλαίσιο. Θα πρέπει να πούμε ότι θέλουμε να συνεχίσουμε τις σχέσεις μας με την ε, χώρα αυτή ε, και στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Η Αίγυπτος είναι πολύ σημαντικός εταίρος, αλλά παίζει και πολύ σημαντικό γεωπολιτικό ρόλο όσον αφορά την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Και ε, επίσης στηρίζουμε τη δημοκρατική μετάβαση στην Αίγυπτο. Επιθυμούμε τον σεβασμό για το κράτος δικαίου και για τις θεμελιώδεις ελευθερίες και δικαιώματα. Και αυτό επιθυμούν και οι ίδιοι οι Πολύ σημαντικά είναι αυτά τα ζητήματα. Έπειτα θα πρέπει να σκεφτούμε προσεκτικά την εφαρμογή του συντάγματος, το οποίο τέθηκε σε ισχύ πριν από ένα χρόνο περίπου. Είναι καλύτερο σύνταγμα από αυτό που ίσχυε στο παρελθόν. Ωστόσο αυτό που τώρα είναι σημαντικό είναι ότι πρέπει να αποτελέσει ε, κομμάτι του θεμελιώδους ε, δικαίου και γι' αυτό είναι σημαντικά τα όσα είπε η κυρία Μογκερίνλα. Θα ήθελα να παροτρύνουμε τους Αιγύπτιους να εφαρμόσουν το Σύνταγμα ε, μετά από τα όσα είδαμε στην τελευταία μας ε, αποστολή παρατήρησης εκεί που, της οποίας ηγήθηκε ο συνάδελφος Μάριο Ντάβιντ. Οι Αιγυπτιακές αρχές θα πρέπει προσεκτικά ε, αλλά και ανοιχτά να προχωρήσουν ε, στα προγραμματά τους. Ευχαριστώ πολύ. Μποστινάρο, παρακαλώ να σέβεστε το χρόνο που σας έχει δοθεί γιατί έχουμε πολύ μεγάλη καθυστέρηση και μετά από αυτή τη μακρά συζήτηση έχουμε ακόμα μία. Κάνω έκκληση στην ευαισθησία σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι. Είναι η μαξιομνημόνευτη αυτή η μέρα. Η είπατε εκπρόσωπος έμεινε στο κοινοβούλιο για πάνω από 7 ώρες. Είναι χειρονομία σεβασμού για το κοινοβούλιο. Ευπρόσδεκτη χειρονομία. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω ρουμανικά τώρα. Το θέμα λοιπόν της Αιγύπτου είναι σημαντικό. Είναι σημαντική χώρα η Αίγυπτος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήδη υπόθηκε και θα πρέπει να υπογραμμιστεί. Πρέπει να θυμόμαστε τον ειδικό ρόλο, τον ιδιαίτερο ρόλο που έπαιξε η Αίγυπτος όσον αφορά τη σύγκρουση στη λωρίδα της Γάζας. Την συνεισφορά που πραγματοποίησε η Αίγυπτος όσον αφορά την αντιμετώπιση των ε, διαφόρων απειλών που την περιβάλλουν. Από αυτή την έποψη η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται ιδιαίτερα όσον αφορά τον εξυγχρονισμό και τον, εκδημοκρατικό, τον εκδημοκρατισμό της ε, Αιγύπτου και των γειτονικών χωρών και ελπίζουμε ότι η Αίγυπτος θα σημειώσει πρόοδο Βεβαίως ανησυχούμε για την παρούσα κατάσταση στην Αίγυπτο όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Κατανοούμε ότι η κατάσταση είναι περίπροκότατη μετά την Επανάσταση στην Αίγυπτο και κατανοούμε και τις μεγάλες τρομοκρατικές απειλές που αντιμετωπίζει η χώρα. Κατανοούμε όλες ιδιαίτερα το θέμα λόγω του πρόσφατου γεγονότος στην, στο Παρίσι και καλωσορίζουμε τις προσπάσεις που καταβάλει ο πρόεδρος Σίση όσον αφορά ε, την προσέγγιση των μουσουλμάνων, την οτροπία των μουσουλμάνων στην Αιγύπτο και καλωσορίζουμε λοιπόν την προσέγγιση αυτή. Αν θέλουμε έναν πιο ήσυχο κόσμο με λιγότερες απειλές είναι σωστή προσέγγιση. Οι κοινοβουλευτικέ εκλογές είναι κάτι που περιμέναμε επί μακρόν. Για τη βελτίωση της δημοκρατίας στην Αίγυπτο ελπίζουμε να είναι ελεύθερη η ψηφοφορία και ελπίζουμε η εκστρατεία να μπορεί να ε, γίνει κανονικά και να συμμετάσχουν όλοι. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αυξήσει τη συνεργασία του με το Κοινοβούλιο της Αιγύπτου, ούτως ώστε να γίνουν οι εξελίξεις που αναμένουμε στην Αιγύπτο. Ο κ. Τάνοκ έχει το λόγο, εκτός μικροφώνου. μετά τον πρόεδρο Μουμπουγάρα έκανε πολλές αλλαγές η Αιγύπτος και υπήρχε μεγάλη αναστάτωση πολιτική. Μετά όταν έφυγε ο πρόεδρος Μόρση κατόπιν επαναστάσεως εναντίον του και τις κατευθύνσεις που ακολουθούσε, τώρα βλέπουμε τις απαρχές σταθερότητας για μια ακόμη φορά, για τη μεγάλη αυτή χώρα. Έκτοτε, υιοθετήθηκε νέο σύνταγμα, μέσω δημοσιοφίσματος. Εξελέγει ο πρόεδρος Αλσίση και πρόσφατα ανακοινώθηκαν βουλευτικές εκλογές. Ευπρόσδεκτα επιτεύγματα. Όμως, είναι η αρχή του ταξιδιού, όχι το τέλος. Πολλά εσωτερικά θέματα πρέπει να ρυθμιστούν αν θέλουμε Αίγυπτος να γίνει πλουραλιστική αραβική δημοκρατία, πολυφωνική δημοκρατία. Το αξίζει και ο λαός της. Η ομάδα μου καλωσορίζει τις βελτιώσεις. Όσον αφορά τους κόπτες χριστιανούς και άλλες μειονότητες, όμως αυτή η ανεξιθρησκεία πρέπει να, να διαπλωθεί, να υπάρχει ελευθερία έκφραση, το δικαίωμα να διαμαρτύρεται κανεί ειρηνικά, το κράτο δικαίου. Είναι βασικά στοιχεία τη δημοκρατία και αυτά επίση θα πρέπει να γίνουν σεβαστά. Πολλοί πολίτε έχουν κατηγορηθεί μέχρι τώρα και φυλακίζονται και έχουν δεχτεί ποινές διότι ασκούσαν αυτά τα δικαιώματα χωρίς βία. Και το γεγονός αυτό δημιουργεί ανησυχίε. Από τον Ιούλιο του 2013 ξέρουμε ότι πάνω από 40.000 ανθρώπους φυλακίστηκαν και 1.400 διαδηλωτές σκοτώθηκαν και αυτά είναι πολύ ανησυχητικά. Και περιορίζεται και ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Η Σου Τάρτον τη εκλογική μου περιφέρεια από δημοσιογράφο τη Αλτζατζίρα δικάστηκε ερήμην και δεν μπορεί να ξαναρχίσει τη δουλειά τη στην περιοχή, να δουλεύει στην περιοχή. Ευρύτερα, μην ξεχνάμε το εξή. Η Αίγυπτο έχει ένα ρόλο. Μπορεί να ηγηθεί του ραβικού κόσμου. Να είναι περιφερειακό φορέα και δύναμη. Μπορεί να παίξει ρόλο για την εξέβρεση λύσεων. Να βελτιωθεί η κατάσταση όσον αφορά τη γειτονική Λιβύη να καταπολεμηθούν οι Ισλαμιστές τρομοκράτες στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική. Σαν φίλος μπορεί να κερδίσουμε πολλά από θετικές σχέσεις με τη μεγάλη χώρα την Αίγυπτο. Είναι πολύ καλό το ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου που θέλει να στηρίξει την Αίγυπτο στη μετάβαση που κάνει στη δημοκρατία. Είναι μεγάλη πρόκληση αυτή η μετάβαση για την χώρα. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Βαν Μπάλεν, έχετε το λόγο. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ίδια η Αιγυπτός δεσμεύτηκε με βάση το νέο της σύνταγμα. Στο νέο της σύνταγμα, αυτό που είναι καλύτερο από το προηγούμενο πιστεύω, τα δικαιώματα του ανθρώπου εντάσσονται στη σωστή θέση, όπως η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Έτσι λοιπόν πρέπει να έρθει στο ύψος των δεσμεύσεων αυτών η Αίγυπτος που ίδια ανέλαβε αυτές τις δεσμεύσεις. Και συμφωνώ με τους προλαλήσαντες ότι εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βρεθούμε στο πλευρό εκείνων που ζητούν την ελευθερία και δημοκρατικά αγωνίζονται για αυτές τις ελευθερίες και που τώρα θα πρέπει να, με βάση τα νομοθετήματα αυτά να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη. Και σε σχέση με τα όσα είπε ο Τσάρλ Στένοκ, η Αίγυπτος θα πρέπει να έχει ένα ζωτικό ρόλο και θα πρέπει να βρει τη θέση της σε αυτό το ρόλο. Μετά τις προεδρικές εκλογές θα γίνουν τώρα οι κοινοβουλευτικές εκλογές και θα ήταν μεγάλο το όφελος αν θα είναι ελεύθερες και δίκαιες αυτές οι εκλογές γιατί είναι ένα περαιτέρω λιθαράκι για την οικοδόμηση της πραγματικής δημοκρατίας και πέρα από την επαγρύπνηση να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την Αίγυπτο να εσέβεται τα δικαιώματα του ανθρώπου με ένα πρόγραμμα γειτονίας ή πατή εκπρόσωπος να δει τι μπορεί να γίνει σε σχέση με τα δικαιώματα του ανθρώπου λοιπόν. Ευχαριστώ. Η κυρία Ματίας παρακαλώ έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Κυρία Αντιπρόεδρε πραγματικά η διάγνωση είναι παρόμοια για την Αίγυπτο. Περνά μια δύσκολη περίοδο και αστάθειας η Αίγυπτος και γι' αυτό τα πράγματα δεν μπορούν να εξετάζονται μόνο στο άσπρο μαύρο. Όλοι γνωρίζουμε ποιες είναι οι απειλές που αντιμετωπίζουν τα δικαιώματα του ανθρώπου, η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία του συναθρίζεσθε όπως αναφέρατε εσείς είπατε εκπρόσωπε. Εμείς πρέπει να μάθουμε από τα μαθήματα του παρελθόντος. Και ιδιαίτερα στα τέσσερα χρόνια που είδαμε, παρακολουθήσαμε αυτή την περιοχή. Είναι αναγκαίο να συναγάγουμε τα μαθήματα από αυτά. Το πρώτο από τα μαθήματα είναι να αποφύγουμε να κάνουμε μαθήματα σε άλλους. Το μέλλον της Αιγύπτου περνά υποχρεωτικά από τα χέρια και τις αποφάσεις των ίδιων των Αιγυπτίων, του λαού της Αιγύπτου. Σε αυτή τη διαδικασία πρέπει και μπορεί να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να βοηθήσει ως διαμεσολαβητής. Διαμεσολαβητής μεταξύ των δύο ε, πλευρών, δύο ε, όχθεων. Και η ε, διοργάνωση των κοινοβουλευτικών εκλογών είναι ένα θετικό βήμα, μια θετική εξέλιξη. Πρέπει να λάβουμε όμως υπόψη ότι η Αιγύπτη είναι υπεύθυνη για όλα αυτά. Έχουμε σίγουρα κοινού στόχους και η κυρία Αντιπρόεδρος πολύ καλά αναφέρθηκε στο ότι πρέπει να βρούμε και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε καλύτερα σε αυτή τη διαδικασία την Αίγυπτο. Και πρέπει τα δικαιώματα αυτά να είναι της Αιγύπτου, των Αιγυπτίων. Οι ίδιοι να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Και για να ολοκληρώσω υπάρχει βαθύτατος σεβασμός ε, σε σχέση με το Ευρωκοινοβούλιο. Είναι μια τιμή να μπορούμε να έχουμε μια τέτοια αντιμετώπιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως αυτή που έχουμε από την κυρία Μογκερίνη. Ευχαριστώ. Σαρτζεντίνη. Σαρτζεντίνη παρακαλώ. Ευχαριστώ. Για τέσσερα ολόκληρα χρόνια οι Αιγύπτιοι βρέθηκαν ε, απελευθερώθηκαν από έναν δικτάτορα, τον δικτάτορα Μουμπάρακ. Το χαιρετήσαμε αυτό εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, χωρίς να σκεφτούμε και να προβληματιστούμε γιατί είχε διατηρηθεί επί τόσα έτη στην εξουσία ο κύριος Μουμπάρακ κατά το παρελθόν. Μετά ακολούθησε ο πρόεδρος Μόση που θεωρήθηκε ότι δεν ήταν απόλυτα δίκαιος και ότι δεν ήταν η δικαιότερη επιλογή και εμείς δεν είμαστε ικανοποιημένοι με το Μόση όμως είχε εκλεγεί και στη συνέχεια απέκτησε ιδιαίτερα δικαιώματα τα οποία έδωσε στον εαυτό του και δεν ικανοποιηθήκαμε καθόλου με αυτή την εξέλιξη είχε αποκλειστικές εξουσίες και αποτέλεσμα ήταν ένα στρατιωτικό πραξικόπημα. Και πολλοί είπαν, ωραία, έγινε ένα στρατιωτικό πραξικόπημα λοιπόν στην Αίγυπτο. Και τώρα τι έχουμε, έχουμε απέναντί μας ένα στρατοκρατικό καθεστώς. Δεν λέω ότι το παρελθόν ήταν καλό, δεν λέω ότι χρειαζόμαστε το Μουμπάρακ ή το Μόση, καθόλου. Όμως αυτά τα οποία βλέπω σε αυτή τη συζήτηση, ο τόνος αυτός μεταξύ των έξι μηνών που ε, πέρασαν από την τελευταία φορά και τώρα λέγοντας ότι είναι τέρος μας στην περιοχή αυτή του κόσμου η Αίγυπτος και πρέπει να βοηθήσουμε για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σίγουρα έγιναν και τα συμβάντα στο Παρίσι όμως όλα αυτά τα βρίσκω εξοργιστικά κυρίες και κύριοι δεν είναι δυνατόν εμείς επειδή φοβόμαστε να και με φοβίες να αντιδρούμε και δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι η Αιγύπτη δεν μπορεί να είναι ελεύθερη και πρέπει να ξανα να βρεθούν υπό στρατιωτικό καθεστώς, υπό μια δικτατορία. Δηλαδή τι, ε, υπό τον Μουμπάρακ ήταν ήσυχοι οι Αιγύπτιοι και βρισκόντουσαν σε μηδενικό σημείο. Οι ε, ακτιβιστές για τα δικαιώματα του ανθρώπου συλλαμβάνονται και καταδικάζονται. Και πρέπει να κατανοήσουμε εμείς ε, στο Ευρωκοινοβούλιο ότι οι ακτιβιστές δεν μπορούν να την χάνουν τέτοια αντιμετώπιση. Ευχαριστώ. Καστάλτο παρακαλώ. Grazie, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Αίγυπτο σήμερα είναι στο μάτι ενός κεκλώνα που συνταράσει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και μεγάλο κομμάτι της ε, Αφρικής. Ε, κράτος δικαίου, ελευθερία έκφρασης, ελευθερία του συνέρχεστε, δικαιώματα απολυτικά και πολιτικά ανάμεσα σε ειλικρινείς ε, φίλους ε, χρέος μας είναι να δείξουμε στον άλλον ε, τον καθρέφτη μπροστά του να αναγνωρίσουμε ωστόσο αντικειμενικά το μεγάλο ρόλο που έχει παίξει η Αίγυπτος στην αντιτρομοκρατική προσπάθεια αλλά και στην επίτευξη ειρήνευσης ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Ωστόσο θα πρέπει να δοθεί προσοχή όσον αφορά τις θρησκευτικές μειονότητες είναι ένα μήνυμα αισιόδοξο, αλλά δεν αρκεί. Ωστόσο, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει στι επόμενε εκλογέ να δούμε ε, και να καλέσουμε σε μια υγιή προσέγγιση more for more, περισσότερα για περισσότερα στη Μεσογειακή Λεκάνη. Αν στου επόμενου μήνε δεν γίνουν αυτά τα βήματα που πρέπει, τότε θα πρέπει να επικρίνουμε με την απαραίτητη ισχύ. Απόψε, ωστόσο, θέλουμε μια μεγάλη και άμεση προσπάθεια, απελευθέρωση δηλαδή των δημοσιογράφων και των bloggers που κρατούνται στη χώρα για να δοθεί αυτό το πνεύμα, αυτός ο αέρας ελευθερίας που ενέπνευσε και την Επανάσταση. Σοπράντ. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένα Ισλάμ το οποίο εντάσσει τις ε, ε, προσταγές του Κορανίου ε, μέσα στο κράτος και δέχεται ότι το, η κρατική αρχή, η κρατική εξουσία είναι ανώτερη από την Σαρία, αλλά υπάρχει και το αντίθετο και αυτό το Ισλάμ είναι το οποίο έχει κηρύξει πόλεμο εναντίον μας. Πρέπει να έχουμε συμμάχους τους μουσουλμάνους. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν αποκλείσει προκλήσει τις ε, κυβερνήσεις ε, που προσπαθούσαν να εντάξουν στο κράτος το Ισλάμ, στο Ιράκ, στη Λιβύη και έδωσαν έφορο έδαφος στους Ισλαμιστές. Ποιο θα είναι το επίπεδο της, ε, της Γαλλίας αν βλέπουμε τι συμβαίνει στην Αίγυπτο. Βλέπουμε πώς πάγωσε το κράτος στη Γαλλία μόνο και μόνο λόγω τριών τρομοκρατών. Ενώ τους τελευταίους 18 μήνες στην Αίγυπτο είχαμε 500 νεκρούς ο Αμπτέλ Φατά έκανε μια έκτακτη εξαιρετική έκκληση. Ζήτησε τα αραβικά κράτη να καθαρίσουν τους, ε, τα ίδια τους ε, ακραίους. Δεν μπορούμε εμείς να δίνουμε διδάγματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Και η ώρα να βρούμε συμμάχους και να αναλάβουμε ε, την ευθύνη των πολιτικών διαφορών που έχουν μαζί μας. Δεν πρόκειται για χειραγώγηση των αισθημάτων, ούτε για παιδεριώδη συνθήματα που περιμένουν οι πολίτες. Θέλουν υπεύθυνα και θαραλέα ε, μηνύματα οι λαοί. Εμείς έχουμε κάνει αυτές τις επιλογές εδώ και χρόνια γιατί η προτεραιότητά μας είναι να ζήσουν ειρηνικά οι λαοί μας και να διατηρήσουν τον πολιτισμό τους. Ο κύριος Γκάμπ, η κυρία Γκάμπριελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Πατεκπρόσωπε, η Αίγυπτο είναι με τι χώρε που θα παίξει αποφασιστικό ρόλο στην απασταθεροποίηση τη περιοχή τη Μεσογείου και όχι μόνο όπως υπενθυμίσατε απλώς. Θα επιμείνω επί πέντε στοιχείων. Πρώτα απ' όλα θα επιμείνω επί της εφαρμογής διαφόρων συνταγματικών διαδικασιών όσον αφορά το δίκαιο και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Ξέρουμε ότι η απαρίθμηση των αρχών και των δικαιωμάτων δεν αρκεί, χρειάζονται συγκεκριμένες δράσεις. Όχι μόνο προεκλογικέ υποσχέσει, θα πρέπει να φροντίσουμε τόσο ώστε οι αρχέ να σεβαστούν πραγματικά το Σύνταγμα. στο το καταφέρουμε αυτό. Δεύτερον, ελευθερία του τύπου και τη έκφραση ή ούτε σταθερότητα ασφάλεια δεν ταιριάζουν με φυλακισμένο τύπο. Αντιθέτως, η ουτε σταθεροτητα ούτε ασφαλεια δεν ταιριαζουν με φυλακισμενο τυπο Αντιθέτω, η ελευθερια των ΜΜΕ θα επιτρέψει να δημιουργηθεί μια πολυφωνική δημοκρατική κοινωνία, διότι εκείνη αποτελεί ένα από τα εργαλεία του διαλόγου εντό τη κοινωνία, Α, τα μέσα επιτρέπουν το διάλογο και ο διάλογο θα αποφύγει την πόλωση τη κοινωνία Αιγύπτου. Τρίτον, πιστεύω ότι ο διάλογος μεταξύ των θρησκειών θα μπορούσε να μειώσει κατά πολύ τι εντάσει και θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη πολυφωνία. ανθαρρύνων την κυβέρνηση Αιγύπτου και την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξουν τι διάφορε πρωτοβουλίε που προωθούν την αμοιβαία κατανόηση και την ανεξιθρησκεία. Τέταρτον, ο ρόλο των γυναικών. Χωρί τη συμμετοχή των γυναικών, η μετάβαση η δημοκρατική δεν μπορεί παρά να είναι μερική. Θα πρέπει να αγγιηθούμε τα δικαιώματά του, να καταπολεμήσουμε τη βία κατά των γυναικών, να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή του όσον αφορά τη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Και εκεί χρειάζονται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες με αποτελέσματα και με τη συμμετοχή των ανδρών και με τη συμμετοχή της Ένωσης. Τέλος, η καταπολέμηση του εμπορίου ανθρώπων είναι μεγάλη πρόκληση και η Αίγυπτος επιτίθεται κατ' του θέματος αυτού και μπορούμε να συνεργαστούμε περαιτέρω. Έχουμε τα μέσα, θα πρέπει τώρα να γίνουν επιχειρησιακά, να λειτουργήσουν, να εφαρμοστούν. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Η υποστήριξή μα θα πρέπει να ανταποκριθεί στο ύψο αυτών, ούτω ώστε να ενισχύσουμε του θεσμού και την Αιγυπτιακή Δημοκρατική Κοινωνία, διότι χωρί αυτού δεν θα υπάρχει βιώσιμη σταθερότητα τη ε, χώρα. Σα ευχαριστώ. Κύριο Χάουιτ έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι σημαντικό εταίρο Ευρωπαϊκή Ένωση η Αίγυπτος, πράγματι αλλά συζητούμε ένα ψήφισμα και το ψήφισμα επικρίνει την Αίγυπτο και θέλουμε να ακουστούν οι επικρίσεις. Ε, υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στη χώρα δέκα 10.000 άνθρωποι του 2004 συνελήφθησαν ε, λόγω σαμποτάζ, τρομοκρατίας ε, και ταραχών και δεν είναι αξιόπιστη δικαιοσύνη και το κατός δικαίου. Μου είπε η Αιγύπτια εκπρόσωπος ότι δεν σωστή στιγμή να διαμαρτύρω για την θανατική ποινή έδωσαν θανατικές ποινές για χιλιάδες υποστηρικτές που έδιωξαν τον Μοχάμεντ Μούρση, τον πρόεδρο. Δεν είναι θέμα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τον πρόεδρο. Διαφωνούμε απόλυτα, κάθετα και πάντα με τις θανατικές ποινές. Η Αίγυπτος πρέπει να καταλάβει ότι με αυτά που κάνει βλάπτεται η εικόνα της η Διότι κρατούνται ακόμα οι δημοσιογράφοι του Αλτζαζίρα. Κανείς εκτός της χώρας δεν πιστεύει ότι είναι κάτι άλλο παρά πραγματικοί δημοσιογράφοι. Και τελικά όταν το νότατο δικαστήριο ανέτρεψε τις κατηγορίες θα πρέπει να απελευθερωθούν. Και η επίθεση κατά των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔ που συνελήφθησαν υποτίθεται 26 ε, ομοφιλόφιλοι. Έχουν αποσυρθεί κατηγορίες κατά αυτών. Πρέπει να γίνονται σεβαστά τα σεξουαλικά δικαιώματα όπως τα άλλα ανθρώπινα δικαιώματα. Τέλος. Ποιο είναι το περιεχόμενο του νόμου για τι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Πρέπει να το εξετάσουμε. Οι διεθνεί οργανώσει και δωρητέ να παίξουν σωστά το ρόλο. Να αρέουν ελεύθερα ιδέε. Χωρί να υπάρχει παρέμβαση από πλευρά κυβερνήσεω κατά του Αιγυπτιακού λαού. Σύμπραξη και συνεργασία σημαίνει πραγματικά σύμπραξη και συνεργασία. Συνάδελφε Δεσμάκερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Χάουιτ, μου κόψατε, μου, πήρατε τα λόγια από το στόμα μου. Ε, Οι ε, δημοσιογράφοι του Αλτζαζίρα βρίσκονται ακόμα στην ε, φυλακή απλά και μόνο επειδή είναι δημοσιογράφοι. Ε, θα πρέπει λοιπόν να τηρούνται και να γίνονται σεβαστές οι πολιτικές ελευθερίες, να μπορεί να γίνει η να υπάρχει μάλλον ε, πολιτική ελευθερία και όλα αυτά υποτίθεται ότι είναι νόμιμα λόγω της καταπολέμησης του τρομοκρατίας και των Ισλαμιστών όμως ε, ο σκοπός δεν αγιάζει κάποτε, πάντοτε τα μέσα γι' αυτό και συμφωνώ κυρία Μογκερίνη να τονίσετε τα θεμελιώδη δικαιώματα και ε, να φροντίσετε για τις εκλογές. Ο κύριο Κουτσούκ, ευχαριστώ. Σήμερα συζητάμε για την κατάσταση στην Αίγυπτο ένα χρόνο μετά από την έγκριση του νέου συντάγματος από τη χώρα αυτή. Το συνταγματικό δημοψήφισμα ήταν ένα σημαντικό βήμα για την δημοκρατία και η Ευρωπαϊκή Ένωση το υποστήριξε. Δυστυχώς οι προεδρικές εκλογές του Ιουνίου δεν έφεραν την σταθερότητα και ένα τμήμα των όσων έμειναν ε, στο κενό ε, και έμειναν μάλλον εκτός των πολιτικών εξελίξεων είναι αυτές που ε, ε, ε, οδηγούν στις παρεκτροπές. Ε, η φυλάκιση φοιτητών και δημοσιογράφων αποσταθεροποιούν τη δημοκρατία. Ωστόσο η Αίγυπτος παίζει πολύ σημαντικό περιφερειακό ρόλο και θα πρέπει να γνωρίσουμε την προσπάθεια για να σπάψουν οι εχθροπαρακτήσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Γάζα, τις προσπάθειες που καταβάλει για το διάλογο στη Λιβύη, για να Υπάρξουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Σουδάν και την Αιθιοπία. Θα πρέπει λοιπόν να μπούμε σε διάλογο με ολόκληρη την Αιγυπτιακή κοινωνία. Κύριος Λεγιαρίκα αυτό που ονομάστηκε άνοιξη αραβική, δηλαδή λαϊκό κίνημα που προσπαθούσε να απελευθερωθεί και να βρει τη δημοκρατία, τελικά δεν είχε πραγματική πολιτική υποστήριξη, πολιτισμική και κοινωνική στήριξη από πλευρά των δικών μα ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Το πνεύμα τη ελευθερία και τη κυριαρχία θα έπρεπε να υποστηριχθεί περισσότερο σε ένα πλαίσιο από εξωτερικέ αναμίξει στην περιφέρεια, όπω η παρέμβαση στη Λιβύη, απελευθέρωσαν τις δυνάμεις της βαρβαρότητας και του φονταμεταλλισμού, η Αίγυπτος ε, γνώρισε πολλές ε, ταραχές και δεν κερδίθηκε η ελευθερία το Αντίθετο, οι μουσουλμάνοι της αντιπολίτευσης του τύπου εκτελέσεις μετά από μαζικές δίκες δεν είναι κάτι αποδεκτό. Θα πρέπει ε, να στηρίξουμε το λαό και να λάβουμε υπόψη την περιφερειακή διάσταση της χώρας. Επί μακρόν ήταν πολιτισμικός φάρος της περιοχής και ήταν ένα στοιχείο που διευκόλυνε το διάλογο, όλος ιδιαίτερος για το διάλογο μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Μια διαδικασία που παρακολουθείτε θα πρέπει να ξεκινήσει στη χώρα, ούτω ώστε να υπάρχει βιώσιμη συνανάπτυξη κάθε πλευρά τη Μεσογείου. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Ζολή. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Ήπατη εκπρόσωπε, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι η πρώτη φορά που συζητούμε εδώ την κατάσταση στην Αίγυπτο. Δυστυχώς, ενώ μερικοί τολμούν να μιλούν ακόμα για μετάβαση δημοκρατική, η κατάσταση συνεχώς επιδεινούται. Η Αίγυπτος έχει πάνω από 15.000 πολιτικούς κρατούμενους. Το 1 τρίτο είναι ακτιβιστές ε, που δεν ανήκουν σε σχετική ομάδα. 147 ε, είναι συνάδελφοί μας. Σαν πρώην δικαστής δεν μπορώ παρά να καταγγείλω την έλλειψη ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος στην Αίγυπτο. Η δικαιοσύνη ούτως υπήν δεν είναι παρά μόνο ένα εργαλείο καταστολής, τυφλής ε, που εφαρμόζεται χωρίς διάκριση από το κράτος εκείνοι που κυβερνούσαν ένα περίπλοκο σύστημα διαφθοράς παλιά ε, αθώθηκαν. Οι νέοι ακτιβιστές όμως από την άλλη πλευρά, η Σάνα Σαΐφ και η Γιάρα Σαλάμ έχουν καταδικαστεί μαζί με άλλους 23 σε δύο χρόνια φυλάκισης. Το μόνο τους έγκλημα είναι ότι διαδήλωσαν για να καταγγείλουν τους νόμους που σκοτώνουν την ελευθερία που θέσπισε το καθεστώς. Η Αίγυπτος θα πρέπει εντάχει να ξαναβρει το μονοπάτι της δημοκρατικής μετάβασης. Διαφορετικά θα πεθάνουν οι ελπίδες που γεννήθηκαν από την Επανάσταση. Συνάδελφε Μπασίρ, έχετε το λόγο. Thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Αίγυπτος κλονίζεται ακόμα από τις επιπτώσεις ε, της Αραβικής Άνοιξης. Βασίζεται ιδιαίτερα στον τουρισμό. Μπορώ ίδιος να ματηρήσω να δώσω τη ματηρία γιατί πήγα εγώ ίδιος εκεί. Η αστάθεια, ο κίνδυνος διώχνουν τους τουρίστες και αυξάνεται η φτώχεια και η απόγνωση. Είναι θλιβερό ότι η βιομηχανία του τουρισμού έχει σήμερα βρίσκεται σε ερήπια μετά από την ε, στρατιωτική δικτατορία που καταδίκασε σε θάνατο εκατοντάδες αδερφούς μουσουλμάνους μεταξύ αυτών όμως και δημοσιογράφους αντιφρονούντες ε, και αθώους διαδηλωτές ε, υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις εδώ και σε σχέση με το Freedom House μια πολύ αξιοσέβαστη οργάνωση με μια έκθεση που δημοσίευσε λέει ότι σε σχέση με την ε, ελευθερία της κοινωνίας βαθμολογείται με πολύ χαμηλό βαθμό παγκόσμια η Αίγυπτος. Μια άλλη πρόκληση σε σχέση με την οργάνωση Open Doors στην έκθεση της αναφέρει ότι δεν υπάρχει θρησκευτική ελευθερία στην Αίγυπτο. Τώρα με απόγνωση ακούμε ότι ο δικτάτορας Χόσνη Μουμπάρακ αθωώθηκε σε σχέση με τις κατηγορίες για τους θανάτους εκατοντάδων διαδηλωτών και την κατάχρηση εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων που χρειάζονται οι πολίτες αυτής της χώρας. Σε σχέση με τους γείτονες είναι, έχει πάρα πολλά προβλήματα και δημιουργεί προβλήματα η Αίγυπτος. Αρνείται τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στα νερά του Νείλου και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ονορεύολε Ομπερμάιερ. Ομπερμάιερ παρακαλώ στη συνέχεια. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ θερμά την κυρία Μογκερίνη και πραγματικά την επενώ για τον χρόνο που μας αφιέρωσε. Κυρίες και κύριοι, το 2014 η Αίγυπτος βελτίωσε την κατάσταση των μειονοτήτων, ιδιαίτερα των χριστιανών. Όμως δυστυχώς μόνο στα χαρτιά η ζωή των κοπτών είναι, συνεχίζει να είναι πάρα πολύ δύσκολη και σε σχέση με την νομική προστασία και την πραγματική προστασία η κατάσταση δεν συγκλίνει. Και βλέπουμε ότι η κατάσταση στην ε, Αίγυπτο υπάρχουν ε, διαρκώς ε, ε, απαγωγές και δολοφονίες και σε άλλους τομείς οι κόπτες υφίστανται αρνητική διακριτική μεταχείριση και η νομοθεσία όσον αφορά την κατάσταση στην εκπαίδευση, την παροχή υπηρεσιών υπάρχει διαρκής αρνητική διάκριση εις βάρος των κοπτών και βλέπουμε εδώ σε σχέση με τον δίκτυ διώξεων βρίσκεται η Αίγυπτος πάρα πολύ χαμηλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιληφθεί των, της προστασίας των μειονοτήτων, ιδιαίτερα των χριστιανικών μειονοτήτων, όπως στην Αίγυπτο των Κοπτών και πρέπει να υπάρξει νομική προστασία υπέρ αυτών και η συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Αιγύπτου πρέπει να εξαρτηθεί από την προστασία αυτής της μειονότητας. Πρέπει να προστατέψουμε αυτή τη μειονότητα. Σας ευχαριστώ. Σμιλιάν Μον παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Μογκερίνη. Η Αίγυπτος για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικός εταίρος ε, στην λεκάνη της Μεσογείου όπως αναφέρθηκε. Παραδοσιακά έχει πρωτοπόρο ρόλο στον ε, κόσμο των αραβικών κρατών. Είναι σημείο αναφοράς ε, στη νότια όχθη της Μεσογείου. Περνά σήμερα μια πολύ δύσκολη περίοδο. Είναι πάρα πολλές οι αντιπαραθέσεις, οι τριβές, οι συγκρούσεις ε, που έχουν πολλαπλασιαστεί και στην Λιβύη και στην ε, σύραξη μεταξύ Αράβων Ισραηλινών, στην κατάσταση στη Λωρίδα της ε, Γάζας και γι' αυτό χρειαζόμαστε μια Αίγυπτο που θα είναι σημαντικός εταίρος στη διεθνή σκηνή και που θα συνεργάζεται μαζί μας για την αναζήτηση λύσεων σε όλες αυτές τις προκλήσεις και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των τζιχαντιστών. Χρειαζόμαστε την Αίγυπτο για να αποκατασταθεί η ειρήνη και η σταθερότητα που διεκδικεί και απαιτεί όλη αυτή η περιοχή συνολικά και μεταξύ των ε, στοιχείων ταυτότητας ε, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει και το κράτος δικαίου, η πλουραλιστική δημοκρατία, ο καταμερισμός των εξουσιών, ε, τα ατομικά δικαιώματα και η ελευθερία από την μη διακριτική μεταχείριση. Για μας είναι οικουμενικές αυτές οι αξίες και θα θέλαμε να τις συμμερίζονται και να τις απολαμβάνουν, να τις απολαύουν όλοι οι Αιγύπτιοι πολίτες. Γίνεται λόγος για δικαιώματα αλλά δυστυχώς δεν υπήρξε η νομοθετική πραγματική εκείνη ανάπτυξη για την υλοποίηση αυτών των δικαιωμάτων. Ενώ υπάρχουν πολλά νομοθετήματα που δεν ευθυγραμμίζονται με τις ε, συνταγματικές επιταγές. Και για τις επόμενες εκλογές κατά τον μήνα Μάρτιο θα έχουμε σημαντικότατο νομοθετικό ρόλο που θα πρέπει να αναλυφθεί. Ελπίζω ότι αυτές οι εκλογές θα γίνουν σε ένα κλίμα διαλόγου και ανοιχτού πνεύματος και θα είναι το δυνατόν πιο ανοιχτέ. Είναι ένα σημαντικό εταίρο τη Ευρωπαϊκής Ένωσης η Αίγυπτος. Πρέπει να την βοηθήσουμε στη μεταβατική περίοδο προς τον εκδημοκρατισμό και τη δημοκρατία προς όφελος όλων των πολιτών της ε, Αιγύπτου που αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα ούτως ή άλλως. Ευχαριστώ. Βάιντεν Χόλτσερ παρακαλώ στη συνέχεια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε σχέση με την ε, Ευρώπη έχει πολύ μεγάλη σημασία η Αίγυπτος και δεν μπορούμε να είμαστε αδιάφοροι για τα όσα συμβαίνουν σε αυτή την πολυπληθή χώρα της Μεσογείου. Φυσικά η σταθερότητα και η προβλεψιμότητα είναι προς όφελος όλων. Και η Αίγυπτος πρέπει να καταβάλει προσπάθειες να αποκατασταθεί η σταθερότητα. Όμως η σταθερότητα πρέπει να οδηγεί προς την αηφορία. Η κυβέρνηση σε μετά από ένα πραξικόπημα ανήρθε στην εξουσία και έχουμε βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα. Κατά το μάλλον ή έχουμε εδώ και τις προσδοκίες ε, που είχαν δημιουργηθεί από την ε, ε, Αραβική Άνοιξη. Πρέπει εδώ να δούμε όλους τους τομείς και τον κύκλο των αδερφών μουσουλμάνων και το τι πρέπει να γίνει το νομοθέτημα του Δεκεμβρίου 2013 που εφημιστικά λέγεται, αναφέρεται δικαίωμα λαϊκών συναθρήσεων και ε, ε, συναντήσεων. Και έχουμε σήμερα την πρακτική εφαρμογή δικαστηρίων που καταδικάζουν όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Όλα αυτά τα μέτρα συνεισφέρουν στο να διαδίδεται, να επεκτείνεται η δυσφορία και να υπάρχει ένα αρνητικό κλίμα το οποίο δεν είναι υπέρ της σταθερότητας η σταθερότητα όλο και περισσότερο κλειδονίζεται. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ε, στο δημοψήφισμα στο οποίο εγκρίθηκε το ε, Σύνταγμα προβλέπει ότι όλες οι διεθνείς συμφωνίες ε, θα πρέπει να είναι σεβαστές και να τηρούνται. Ευχαριστώ. παρακαλώ στη συνέχεια. E, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή όλων στην κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά τους κόπτες χριστιανούς που είναι 10% του πληθυσμού της Αιγύπτου. Είναι η μεγαλύτερη χριστιανική μειονότητα στη Μέση Ανατολή. Στο Κάιρο τους τελευταίους μήνες αρκετές εκκλησίες, σχολεία και σπίτια κοπτών δέχτηκαν επιθέσεις. Οι κόπτες δεν έχουν πρόσβαση σε υψηλές θέσεις στη δίκηση ή στο στρατό Επίσης, τα καταστήματα των κοπτών σημαδεύονται με, το, με ένα σημάδι, με ένα χ. Οι αρχές δυστυχώς δεν μπορούν να παράσχουν προστασία. Τον Σεπτέμβριο του 2013 ένα χωριό κοπτών υπέστη λαιλασία και ε, ξυλοκόπησαν κόπτες. Δεν ήταν η μουσουλμανική αδελφότητα που το έκανε αυτό. δεν ξέρουν ποιο το έκαναν και έπρεπε οι αρχές κανονικά να κινητοποιηθούν. Μάλλον το Ισλαμικό κράτος ήταν το ενοχό και η, και η διοίκηση τελικά ουσιαστικά φέρνει σε δυσχερή θέση τους κόπτες. Θα έπρεπε να προστατεύονται τα δικαιώματα των χριστιανών, των κοπτών χριστιανών. Κυρία Αντιπρόεδρε, κάτι πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ, επόμενο ομιλητή. Ο κ. Μπόλαν, κυρία Μογκερίνη, σωστά λέει ο κ. Βάγκελ, συγγνώμη, σωστά είπατε στην εισαγωγή σα ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της σημασίας που έχει η Αίγυπτος σαν χώρα, σημασία που έχει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την ειρήνη και τη σταθερότητα στη χώρα, αυτό από τη μια, και από την άλλη πρέπει να δούμε ποιες είναι οι προσδοκίες μας όσον αφορά την Αίγυπτο. Δεν μπορούμε να παραιτηθούμε των προσδοκιών μας όσον αφορά το κράτος δικαίου, ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ατομικά και συλλογικά. Όταν όμως συντάσσουμε ψηφίσματα, θα έλεγα ότι πρέπει να προσέχουμε τον τόνο. Είναι κάπως σκληρό το έγγραφο που ετοίμασαμε. Δεν νομίζω ότι αξίζει τέτοιο τόνο ο Αίγυπτος τώρα. Όταν συντάσσουμε λοιπόν τα ψηφίσματα, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι μια χώρα όπως είναι η Αίγυπτος είναι ένας εταίρος. Εταίρος που χρειαζόμαστε μέσα στην όλη αναταραχή που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Πρέπει να εκτιμήσουμε τι δυναμικό εμπεριέχει αυτή η χώρα, τι δυνατότητες έχει για τη σταθερότητα, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην περιοχή και για, άλλα, για την προστασία στατηγικών συμφερόντων της Υπήρου μας που να παίξει ρόλο. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι σωστό να περιμένουμε από την Αίγυπτο να μετατραπεί σε μια δημοκρατία, να αναπτύξει τους θεσμούς της και να διεξαχθούν δημοκρατικές εκλογές. Σας ευχαριστώ, συνάδελφε Μπόιλαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούσαμε χθε ότι ο Υπουργό Εξωτερικών τη Αιγύπτου είπε ότι υπάρχει μια πιθανότητα ότι οι δημοσιογράφοι τη Αλτζαζίρα ε, να παραχθούν των κατηγοριών. Και θα πρέπει και τον Έμπραμ Αλάου, να τον λάβουμε υπόψη, που είναι έφηβος Ιρλανδός, που ε, κρατείται από τον Αύγουστο 2013 ανευθυντικής. Ο Αμπραάμ στα 17 ήταν παιδί όταν συνελήφθη για πρώτη φορά μετά τις διαμαρτυρίες στο Κάιρο. Έκτοτε θεωρείται ε, κρατούμενο συνείδησης ε, από την Διεθνή Αμναστία. Δεν ε, είχε πληγωθεί στο χέρι από πυροβολισμό και δεν, ε, δεν τον περιέθαψαν κανονικά και έχει πάρα πολύ πρόβλημα, έχει ξυλοκοπηθεί άγρια, είναι στην απομόνωση στη φυλακή, αναβλήθηκε τρεις φορές η δίκη του και σήμερα εξακολουθεί να αντιμετωπίσει μαζική δίκη μαζί με άλλους 493 κατούμενους μαζί με τους οποίους ε, κατηγορείται ελήψη όμως στοιχείων. Δράτω με τις ευκαιρίες να επενθυμίσω στην ύπατη εκπρόσωπο το αίτημά μου να συναντηθούμε, να συζητήσουμε το θέμα του Αμπραάμ το Αβραάμ και να απελευθερωθεί ανεφόρον από την φυλακή. Συνάδελφε Σμιθ. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Συνάδελφοι, όλοι συμφωνούμε ότι η Αίγυπτος είναι ζωτικό στρατηγικό εταίρο στην περιοχή. Συμφωνούμε επίσης, όπως λέμε και στο ψήφισμά μας, ότι η Αίγυπτος έχει με πολύ δρόμο να ακολουθήσει για να φτάσει στις προδιαγραφέ που έχουμε θέσει και έχουμε καθήκον έναντι του Αιγυπτιακού λαού να παρουσιάζουμε τα κενά που έχει η κυβέρνησή τους διότι ήταν τόσο ενθουσιώδης η Αιγύπτη στην Αραβική Άνοιξη και Επανάσταση τελικά δεν θα πρέπει να τις απογοητεύσει. Κυρία Μογκερίνη, εντυπωσιάστηκα με τα σχόλιά σας όπως πάντα. Νομίζω ότι έχουμε κοινό πρόγραμμα μαζί και ελπίζω ότι θα πρέπει να σας ε, στηρίξουμε στις συνομιλίες στις Αιγυπτιακές Αρχές. Ε, αναφέρθηκαν πολιτικοί κρατούμενοι, ε, ΛΟΑΔ, ε, τι μη κυβερνητικέ οργανώσει, δημοσιογράφοι. Είναι σε πολύ επικίνδυνε οι μη κυβερνητικέ οργανώσει στην Αίγυπτο, αλλά στην παράγραφο 17 ζητούμε από την Αίγυπτο να συνεργαστεί με όλου του φορεί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το ΙΕ και άλλου φορεί. Στην παράγραφο 6 λέμε κάτι παραπάνω. Καλούμε την Αίγυπτο να επικυρώσει το καταστατικό για του Ρωμά και ε, της Ρώμης συγγνώμη, και να, επίσης να υπογράψει να γίνει μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Νομίζω ότι θα πρέπει να τους ενθαρρύνουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Αξίζει τον κόπο. Ο κύριος Επιτίδιος έχει το λόγο. Η απειλή η οποία προέρχεται από την τρομοκρατική δραστηριότητα των ε, τζιχαντιστών είναι πολύπλευρη και πολυδιάστατη. Οι ομάδες που πραγματοποιούν τις ε, τρομοκρατικές επιθέσεις στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις δεν είναι μόνο κάτοικοι των πόλεων αυτών έχουν συνεργάτε και ομοειδιάτε στι γειτονικέ μουσουλμανικέ χώρε κυρίω τη νότια γειτονιά τη ευρώπη. εάν επιθυμούμε να περιορίσουμε ή να εξαλείψουμε το φαινόμενο αυτό θα πρέπει να βοηθήσουμε τι κυβερνήσει των χωρών αυτών να απαλλαγούν από του τζιχαντιστέ στη χώρα του ώστε να μην μπορούν αυτοί να έρχονται στην ευρώπη. για να το επιτύχουμε αυτό θα πρέπει να του ε, βοηθήσουμε να βρουν τη χρυσή τομή ανάμεσα στην ε, ασφάλεια και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μία από τις χώρες για τις οποίες η τζιχαντιστική ε, τρομοκρατία αποτελεί απειλή είναι η αίγυπτος. εκεί οι τζιχαντιστές δολοφονούν κάνουν απαγωγές και στοχοποιούν χριστιανούς ιερωμένους κυρίως τους ελληνοορθόδοξους ε, μοναχούς των μονών του όρου σινά. γι' αυτό και το κράτος αντιμετωπίζει τόσο με νομοθετικά μέσα όσο και με στρατιωτικά μέσα. στο σύνταγμα προβλέπεται να είναι εγκλήματα η τρομοκρατία και η διακίνηση των ατόμων. συνεπώς η συνεργασία της ευρωπαϊκής Ένωσης με την αίγυπτο θα συμβάλει στο να αντιμετωπιστεί η τρομοκρατία εκεί και να αισθανόμαστε περισσότερο ασφαλείς εμείς στην ευρώπη. ευχαριστώ. gospodine predsjedniče, jasno je da europska unija mora stabilnost η ευρωπαϊκή ένωση θα πρέπει να υποστηρίξει τη σταθερότητα της στην αίγυπτο και να προαγάγει τις δημοκρατικές εξελίξεις, τον εκδημοκρατισμό αυτής της χώρας. Είναι συμπληρωματική αυτή η δράση. Πρέπει να βοηθήσουμε στην ανοικοδόμηση δημοκρατικών θεσμών και θεσμικών οργάνων, να βοηθήσουμε στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας που πρέπει να είναι προτεραιότητα. Ιδιαίτερα αν εξετάσουμε αυτό υπό το πρίσμα της στρατηγικής συνεργασίας που πρέπει να επιτευχθεί. Η ριζοσπαστική δράση και η τρομοκρατία είναι οι κύριε απειλέ για την ανάπτυξη τη Αιγύπτου. Βραχυπρόθεσμα προτεραιότητα πρέπει να είναι η σταθερότητα στην Αίγυπτο, επειδή η σταθερότητα στην Αίγυπτο έχει στρατηγική σπουδαιότητα για την Ευρώπη. Και θα πρέπει να διασφαλίσουμε μια ευρύτερη ζώνη ασφάλειας και σταθερότητας σε αυτή την περιοχή του κόσμου, σε αυτή την περιφέρεια. Φυσικά υπάρχουν δημοκρατικές ελλείψεις και κενά και χάσματα στην Αίγυπτο. Ευχαριστώ. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη Κυρία Μογκερίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ότι αναφέρατε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όσον αφορά τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου στην Αίγυπτο. Πρόσφατα επισκέφθηκα την Αίγυπτο, μίλησα με τα κόμματα, με τα μέσα και με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και δεξαμενών σκέψεων. Είναι σημαντικό ότι πρέπει τη δημοκρατία, την ελευθερία της έκφρασης, τα θεμελιώδη δικαιώματα να τα πάρουμε πολύ σοβαρά. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι η καταπίεση του καθεστώτος του στρατηγού Σίση της κοινωνίας των πολιτών καταπίεσης με τέτοιο έντονο τρόπο των δημοκρατικών δικαιωμάτων που δεν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα αυτά και να εκφραστούν ελεύθερα οι πολίτες και βρίσκονται στις φυλακές κρατούμενοι. Πρέπει να βοηθήσουμε λοιπόν, να συνδράμουμε. Βρίσκουμε, βλέπουμε μια κατάσταση όπου η Αραβική Άνοιξη και η οδός προς την, τον εκδημοκρατισμό δημιουργεί μια νέα ε, γενεά στρατιωτικού καθεστώτος ε, στρατοκρατών. Φοβούνται οι άνθρωποι ότι θα είναι χειρότερο αυτό το καθεστώς από το καθεστώς του Μουμπάρακ. Πρέπει να γίνουν αλλαγές στον ποινικό κώδικα, ώστε να μην μπορεί να καταδικάζεται κανείς ε, ισόβια επειδή δίνεται διεθνής βοήθεια σε κάποιο όργανο στην Αίγυπτο. Ευχαριστώ. Ζάχαρη στη συνέχεια. Ζάχραντιλ. Ευχαριστώ κυρία Μογκερίνη η κυβέρνηση του στρατηγού Προέδρου Σίση πόρο απέχει από το να είναι μια ιδανική κυβέρνηση για την Αίγυπτο. Από την άλλη πλευρά είναι μια κυβέρνηση αυτή που έχει οδηγήσει σε οικονομική ε, κατάπτωση στην Αίγυπτο. Δείχνεται ότι ε, οι χώρες της ε, του Μαγκρέμπ έχουν δύο δυνατότητες ή τη δυνατότητα ε, ισχυρών καθεστώτων με δικτατορικά χαρακτηριστικά, με δικτατορικά χαρακτηριστικά όπως ε, για παράδειγμα του στρατηγού Σίση ή ενός ιδεολογικού Ισλάμ όπως αυτό το βλέπουμε στην Τινησία, στο Μαρόκο και αλλού. Και το καλύτερο παράδειγμα γι' αυτό είναι η Τουρκία κατά τα άλλα. Φυσικά η δεύτερη οδός είναι καλύτερη από την πρώτη των δικτατορικών καθεστώτων. Όμως πρέπει ως Ευρωπαίοι να συνηθίσουμε την ιδέα ότι καμία από αυτές τις δύο πορείες δεν μπορεί να εγκαθιδρύσει ένα δημοκρατικό καθεστώς σαν αυτό το οποίο θα επιθυμούσαμε εμείς οι Ευρωπαίοι. Μεταξύ αυτών των δύο οδών είναι καλύτερη η πορεία από ό,τι σε σχέση με το Ιράκ ή τη Συρία. Πρέπει με πραγματιστικό, ρεαλιστικό τρόπο να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα και ελπίζω ότι η κυρία Μογκερίνη που ασχολήθηκε με αυτό το θέμα θα καταφέρει να λύσει αυτή, αυτό το πρόβλημα. Λόπετ Μπερμέχο παρακαλώ στη συνέχεια. Εκατομμύρια Αιγυπτίων πήγαν στην πλατεία Ταχρήρ και σε όλες τις πλατείες διεκδικώντας κοινωνικά δικαιώματα και ελευθερίες. Τέσσερα χρόνια μετά βλέπουμε ένα νέο κύμα καταπίεσης σε αυτή τη χώρα με πάνω από 800 νεκρούς ε, και καταπίεση, καταδίκες σε θάνατο, ε, φυλάκιση των ε, αντιφρονούντων, της αντιπολίτευσης των φοιτητών, δημοσιογράφων και βλέπουμε επίσης καταπίεση όσον αφορά τις σεξουαλικές επιλογές. Έχουμε εδώ την ε, ε, τοποθέτηση του στρατηγού ε, Σίση και και την προσπάθεια να ε, καταδικαστεί η σφαγή των ε, Παλαιστινίων από τους Ισραηλινούς. Ε, και σε σχέση με αυτό το οποίο γίνεται στη λωρίδα της Γάζας για την φυλάκιση των ίδιων των κατοίκων της λωρίδας της Γάζας σε μια ανοιχτή φυλακή, όμως το, ο στρατός της Αιγύπτου παίρνει χρηματοδότηση από την Αμερική. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δίνει υποστήριξη σε αυτή τη χώρα χώρα. Το ίδιο έγινε και στο παρελθόν όμως. Δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται η ιστορία. Το μέλλον της Αιγύπτου πρέπει να βρεθεί στα χέρια των Αιγυπτίων πολιτών, χωρίς εξωτερικές αναμίξεις. Και αυτή η ανάμιξη δεν μπορεί να γίνεται ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Μπίκνερ παρακαλώ στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμε είπατε εκπρόσωπε στην Αίγυπτο αυτή τη στιγμή τα δικαιώματα του ανθρώπου κατάφορα ποδοπατούνται και γι' αυτό θα ψηφίσουμε αύριο και θα υπερψηφίσουμε το ψήφισμα εμείς αύριο. Αλλά αυτό μόνο του δεν επαρκεί. Η κατάσταση έχει ως εξή. Οι αδερφοί μουσουλμάνοι με κάθε τρόπο προσπαθούν να επιστρέψουν στην κυβέρνηση. Κάνουν ένοπλες ε, διαδηλώσεις ε, ε, με τις απαγωγές πολιτών δρούν επιθετικά. Σημαντικό είναι ότι μεγάλο μέρος των Αιγυπτίων λιμοκτονεί. Είναι η ευκαιρία αυτή των αδερφών μουσουλμάνων δίνουν μια κάποια βοήθεια σε αυτούς τους λιμοκτονούντες και την χάνουν της υποστήριξής τους. Γι' αυτό έντονη παράκληση. Δεν πρέπει να παραμείνουμε σε αυτό το ψήφισμα μόνο γιατί δεν θα καταφέρουμε τίποτα κατά τα άλλα αν το κάνουμε αυτό. Πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι λόγοι, τα αίτια αυτών των ε, ε, προβλημάτων και πρέπει να αυξήσουμε τη βοήθεια προς την κυβέρνηση ώστε η οικονομία να μπορέσει να ανακάμψει. Γι' αυτό επίγουσα, κατεπίγουσα έκκληση σε εσάς κυρία Ήπατη εκπρόσωπε να αυξηθούν τα κονδύλια στείλει αυτά προς την Αίγυπτο ώστε να μπορέσει η οικονομία της Αιγύπτου να ανακάμψει με αυτή τη βοήθεια. Ευχαριστώ. Νεβουέτα παρακαλώ στη συνέχεια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα πρέπει να πούμε εδώ, Είπατε οι εκπρόσωποι. Ε, ε, ότι αυθαίρετες φυλακίσεις και διώξεις ε, συμβαίνουν στην Αίγυπτο. Υπάρχουν φρικτές περιπτώσεις βασανιστήριων σε σχέση με τους οπαδούς εις βάρος των οπαδών του Προέδρου Μόση. Συλλαμβάνονται χωρίς, καμία, χωρίς ένταλμα οι δικαστικές αποφάσεις και βρίσκονται εδώ, βλέπουμε ότι υπάρχουν καταδίκες που πολιτικά έχουν πολιτικά εμπνευστεί και δημιουργηθεί και βλέπουμε ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις ε, οι δικηγόροι δεν είχαν δυνατότητα να ασκήσουν τα δικαιώματά τους υπέρ των κατηγορουμένων. Μάρτυρες δεν μπόρεσαν να καταθέσουν. Η Αιγυπτιακή δικαιοσύνη δείχνει ότι αυτή είναι μια φρικτή κατάσταση και δεν μπορούν τα πράγματα, δεν λειτουργεί σωστά. Υπήρξαν υποσχέσεις ε, για ένα κράτος δικαίου, όμως υπήρξαν τεράστιες παραβιάσεις και παραβάσεις του κράτους δικαίου και βλέπουμε ότι υπάρχει εντύπωση ότι εδώ ατιμωρητοί μπορούν κάποιοι να παραβαίνουν τον νόμο και ποδοπατούν κατάφορα τον νόμο και την ε, δικαιοσύνη ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι ε, παρατηρητής. Πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να υπάρξει μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη στην Αίγυπτο. Και όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων να προσαχθούν στη δικαιοσύνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει φτάσει σε ανησυχητικά επίπεδα ε, υπό την ε, στρατηγό Σίση. Έχει ο στρατηγό Σίση ε, επιδεινώσει τη δημοκρατική κατάσταση της χώρας του και το συνεχίζει καθημερινά. Οι περισσότερες πολιτικές του δεν θα καταλέξουν σε περισσότερε εξάρσεις του ISIS τα όσα συμβαίνουν εκεί επηρεάζουν ολόκληρη την περιοχή. παράνομε δολοφονίε, φυλακίσεις, δημοσιογράφων, ιδιαίτερα η υπόθεση των τριών δημοσιογράφων του Αλτζαζίρα που πρέπει να απεφεθούν ελεύθεροι άμεσα. Ε, καθημερινά προσπαθούν να πνίξουν την κοινωνία των πολιτών και δεν ε, ε, χρησιμοποιούμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να τα σταματήσουμε αυτό. Θα πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι με τους κρατούμενους και την κοινωνία των πολιτών στην Αίγυπτο. μια ρεαλιστική και δημοκρατική κοινωνία μπορεί να εξασφαλίσει μια μακροχρόνια σταθερότητα και ευημερία στην Αίγυπτο. Ευχαριστώ. Уважаеми господин госпожо Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε. Η κατάσταση στην Αίγυπτο παραμένει πολύ ανησυχητική. Μετά από το κύμα της ε, ε, επανάστασης που έγινε γνωστό ως Αραβική Άνοιξη η, δυστυχώς υπήρξε μια μετατροπή, μια μεταμόρφωση σε ένα μακρύ Ισλαμιστικό χειμώνα οι αδερφοί Μουσουλμάνη είναι μία από τις Ισλαμιστικές οργανώσεις, έχουν επαφές με τους και δεσμούς με τις ένοπλες Ισλαμιστικές δυνάμεις και είναι μεγάλη απειλή για την, περιοχή. για την περιοχή. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, ε, πολλοί ε, Ορθόδοξοι ε, διώχθηκαν. Οι χριστιανοί ακόμα κινδυνεύουν. Εάν οι αδερφοί μουσουλμάνοι είναι τμήμα της εξουσίας στην Αίγυπτο, θα αποτελέσουν μεγάλη απειλή και κατά της Ευρώπης κοντά στην Χαμάς, την Μπόκο Χαράμ, την Αλγάιντα, ε, την Μπόκο Χαράμ και άλλους. Ε, δεν θα πρέπει να υπάρξει δεν υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στους αδερφούς ε, μουσουλμάνους και την κυβέρνηση Ερντογάν στην Τουρκία. Ε, α, τι κάνουμε εμείς για να μπορέσουμε να αντισταθούμε σε αυτή την κατάσταση. Ο κύριος Βέγκας, σε τέσσερα χρόνια απογοητεύσεων με φοβερές φρικαλαιότητες που γίνονται κατά του πληθυσμού. Έχουμε στην ουσία μπροστά μας αυτούς που ποτέ δεν έπαψαν να κυβερνούν στην Αίγυπτο. Γιατί οι ένοπλες δυνάμεις στην Αίγυπτο είναι η πιο ισχυρή εξουσία της χώρας και ο πρόεδρος της το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Η, 1,8 ε, δις δε δίνουν οι ΙΠΑ ε, ετησίως στην Αμερική. Μόνο το Ισραήλ και η Κολομβία ε, παίρνουν περισσότερα από τις ΗΠΑ. Ωστόσο δεν υπάρχει περισσότερη δημοκρατία και κοινωνικά δικαιώματα. Εμείς κάνουμε έκκληση να μπορέσει ο λαός επιτέλους να αποφασίσει για το μέλλον του, να ξεπεράσει τις τοπικές ολιγαρχίες και να άσχετα από τις, τα γεωπολιτικά συμφέροντα της Δύσης. Γκαμπούς παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αντιπρόεδρε, τον Ιανουάριο 2012 μια λαϊκή επανάσταση ανέτρεψε το Μουμπάρακ και προσθέθηκε και η Αίγυπτος στην Αραβική Άνοιξη. Μία ε, άνοιξη όμως που άρχισαν να επιδεινώνονται τα πράγματα. Η κοινωνία της Αιγύπτου ήταν περίπλοκη ήδη κατά την περίοδο του Μουμπάρακ, περίπλοκη κατά την περίοδο Μούρση και περίπλοκη κατά την περίοδο Σίση. Αυτή η περιπλοκότητα είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας κάνει να αναγνωρίσουμε έναν εταίρο, ένα σύμμαχο στην ε, Αίγυπτο. Για τους στόχους ε, της στην ε, Μέση Ανατολή. Αυτό σημαίνει ότι σε συγκεκριμένα μέτρη που ε, έχουν ε, ληφθεί σε σχέση με τα δικαιώματα του ανθρώπου θα πρέπει να υψώσουμε τη φωνή για να υπάρξει επανόρθωση και επιστροφή στο κράτος δικαίου. Και θα πρέπει να μπορέσουμε να τα πούμε αυτά ανοιχτά όπως μιλάνε οι φίλοι μεταξύ τους αλλά και με κατανόηση ότι ο φίλος συνεχίζει να είναι φίλος και καλύτερος φίλος ακόμα και με το πρόγραμμα γειτονίας πρέπει να αποκτήσει σάρκα και οστά και να είναι αποτελεσματικό. Κατανοούμε την ανησυχία του Κοινοβουλίου για τα συμβαίνοντα στην Αίγυπτο και τα συμπτώματα για την βελτίωση και έχουμε τι εκλογέ του Ματίου σαν μια ευκαιρία που αναδύεται. Έχω αμφιβολίες για την ανάγκη ενό τρίτου ψηφίσματο κατά τη διάρκεια διαστήματο μικρότερου από ενό έτος, για την Αίγυπτο. Πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί, πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται ώστε να είναι πραγματική δημοκρατία η Αίγυπτο. Όπω όπως είναι φυσικό για όλα τα μέρη του κόσμου πρέπει να το κάνουμε αυτό. Αλλά να το κάνουμε χωρίς να βλάψουμε αυτό το μεγάλο κινητήρα ισορροπιών που είναι η Αίγυπτο σε αυτή την περιοχή του κόσμου. Ευχαριστώ. Παντσέρι παρακαλώ στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Ξέρουμε όλοι ότι η Αίγυπτος είναι μια χώρα κλειδί στην περιοχή που έπαιξε και που απέξει σημαντικό ρόλο οι γειτονία τη αιστεία του Ισλαμικού κράτου την κάνουν πολύ ευαίσθητη θέση τη εν λόγω χώρας και πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι πρέπει να υπάρχει σωστή ε, προσέγγιση και ισορροπία για την πολιτική θέση. Λοιπόν, αναφεσβήτητα πρέπει να πω ότι είναι αποφασιστική σημασία να ολοκληρωθεί η μετάβαση δημοκρατική στην Αίγυπτο. Διότι είναι η καλύτερη απάντηση που μπορεί να δοθεί σημερινά προβλήματα, κυρίω αυτά που δημιουργούνται από την τρομοκρατία. Και δεν θέλουμε να περιορίσουμε όμω, περιορίζονται οι ελευθερίε στα δικαιώματα. Αντίθετα, να παγιωθεί η δημοκρατία και τα δικαιώματα. Ε, Θεωρούμε σημαντική λοιπόν την Αίγυπτο στο περιφερειακό πλαίσιο. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια Αίγυπτο που θα ενστερνιστεί τις δημοκρατικές αρχές για τις μελλοντικές τρεις δράσεις. Συνάδελφε Ρούας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι σημαντική, σημαντικός ο ρόλος της Αιγύπτου και παρακολουθούμε με ανησυχία την κατάσταση σε αυτή τη χώρα από αυτό το κοσμικό κράτος που απορρέουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τα όσα έχουν συμβεί. Και μάλιστα υπάρχει ανεργία των νέων, ανεργία των γυναικών, υπάρχει φτώχεια, υπάρχει αγραμματοσύνη, είναι μεγάλος ο αναλφαβητισμός και εδώ υπάρχει και η ανησυχία της διεθνούς κοινότητας για την δημοκρατία και την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου εκεί. Με όλα αυτά και παρόλο αυτό το σενάριο στρεφόμαστε με ελπίδες προς το μέλλον, για το μέλλον της Αιγύπτου. Θα γίνουν εκλογές κοινοβουλευτικές που είναι πάντα μια θετική στιγμή για να ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας για αυτή τη χώρα και με ένα σενάριο σταθερότητας, πολιτικής σταθερότητας. Αυτό αναμένουμε και ευελπιστούμε ότι θα γίνει. Μια ανάκαμψη οικονομική που μπορεί να δώσει τη δυνατότητα να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη στην Αίγυπτο. Αναμένουμε τώρα να σέβονται αυστηρά τις οικουμενικές αρχές ε, για τα δικαιώματα του ανθρώπου οι, οι κυβερνήσεις, οι αρχές της Αιγύπτου και αναμένουμε από την ύπατη εκπρόσωπο να παρακολουθήσει αυτές τις εκλογές εκ του σύνεγγης με ιδιαίτερη προσοχή. Ευχαριστώ. Ρορε Γκόμες. Γκόμες παρακαλώ. Η κυρία Γκόμες. Η Αιγυπτιακή ηγεσία έχει να κάνει μια επιλογή ε, θέλει να μπει ε, μέσα στη διεθνή κοινότητα και να μπορέσει να παίξει το ρόλο που της αρμόζει στην Αφρική και στην, ε, στην λεκάνη της Μεσογείου ή θέλει να είναι ένα αυταρχικό κράτος το οποίο καταδικάζει τις πολιτικές ελευθερίες, καταπατά τα βασικά δικαιώματα ενώ απελευθερώνει και αθωώνει τον Μουμπάρακ. Αυτά τα βασικά δικαιώματα ε, δεν ισχύουν. Είναι πραγματικά χονδροειδής η καταπάτησή τους και η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί ανεξάρτητα στην Μεσόγειο. Θα χρειαζόμασταν πολύ μια ε, ισχυρή, ε, αξιόπιστη Αίγυπτο. Αλλά αυτό δεν γίνεται με το στραγγαλισμό της δημοκρατίας. Αντίθετα, ο κάθε Μουμπάρακ κατασκευάζει έναν Μόρση. Η ευρωπαϊκή επιλογή είναι περισσότερο και περισσότερο, μόρφο for Υπάρχει και το αντίθετο, λιγότερο και λιγότερο. Θα χάναμε όλοι στη Μεσόγειο αν από το μεγαλείο των Φαραώ και από την ελπίδα που γεννήθηκε στην πλατεία Ταχρήρε αφήσουμε την Αίγυπτο να καταστραφεί και να πνιγεί, να πνιγεί από τον πρόεδρο ε, Σίση. Έχει τεράστιο δημοκρατικό έλλειμμα στην Αίγυπτο, μια χώρα που διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη Μεσόγειο και στον αραβικό κόσμο και συνιστά εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα η Αίγυπτος δίνει τη μάχη μαζί με τη Δύση ενάντια στην τρομοκρατία και μπορεί να αποτελέσει σταθεροποιητικό παράγοντα της περιοχής μαζί με την Κύπρο, το Ισραήλ και την Ελλάδα αποτελεί σημαντικό εταίρο σε ζητήματα ασφάλεια και ανάπτυξη, ειδικά σε μια περίοδο όπου οι πολιτικέ επενδύσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην δικτατορική τουρκία του Ερτογάν καταραίουν. από κοινού οι χώρε τη ανατολική μεσογείου μπορούν να αποτελέσουν πηγή ενέργεια για την ευρωπαϊκή ένωση συνεπώς η στενή συνεργασία της ευρωπαϊκής ένωσης με την αίγυπτο χαλά τους σχεδιασμούς των φανατικών ισλαμιστών ειδικά μέσα από την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και των θρησκευτικών ελευθεριών όπως και η έκθεση μας εισηγείται. να μην ξεχνάμε ότι κανείς δεν είναι τέλειος και ακόμη και μέσα στην ευρωπαϊκή ένωση έχουμε δημοκρατικά ελλείμματα αλλά η αίγυπτος χρειάζεται τη στήριξη και την ενίσχυση τη Ευρωπαϊκή ένωσης για να αναπτύξει την δημοκρατία της και να την κάνει καλύτερη. Η σταθερότητα στη χώρα θα συμβάλλει στη βελτίωση της δημοκρατίας, στην ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, στη σταθερότητα της περιοχής. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως ήδη ακούσαμε απόψε, ε, το δικαστήριο της Αιγύπτου ανέτρεψε την μόνη καταδίκη που απέμενε κατά του πρώην Προέδρου Μουμπάρακ. Οι πρώτες κατηγορίες για φόνους ε, διαδηλατών και αυτές αποσύρθηκαν. Τέσσερα χρόνια σκληρών θυσιών του Αιγυπτιακού λαού τελικά εις απεδείχθησαν. Έτσι δε περαιτέρω, διότι υπό τον πρόεδρο Σίση εκατοντάδε καταδικάστηκαν στο θάνατο σε μαζικέ δίκε. Ακτιβιστέ τιμωρούνται για ειρηνικέ διαδηλώσει και μη κυβερνητικέ οργανώσει αντιμετωπίζουν μεγάλη καταστολή. Τον Αύγουστο του 2013 περίπου χίλιοι διαδηλωτέ δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν σε εκδηλώσει που δεν είχαν σχέση, που αντιστοιχούσαν με αυτά που είναι στη Διανανμέν. Αντίθετα από την Διανανμέν, ε, ε, δεν ξέρουμε εκείνου που ήταν οι ένοχοι. Οπότε έτσι ρίχνουμε πολλούς αγκαλιές των τρομοκρατικών οργανώσεων. Αν δεν κινηθούμε, τελικά θα είναι επιβλαβές για τους Αιγυπτίους και για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ζητώ την να μας πει η είπατε εκπρόσωπος ποια είναι η στρατηγική σας επ' αυτού δοθέντως ότι η δυτική τεχνολογία και ο εξοπλισμός δίνουν δυνατότητες στις αρχές να καταστέλουν τις κινήσεις των πολιτών. Πρώτο βήμα θα ήταν μήπως πρέπει να απαγορεύσουμε τις εξαγωγές τέτοιων προϊόντων προς την Αίγυπτο και προς ε, παρόμοιες χώρες. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Μακοβέη. Σας ευχαριστώ πολύ. Τον τελευταίο χρόνο στην Αίγυπτο πάνω από 16.000 άνθρωποι συνελήφθησαν, ακόμα και άνθρωποι που βγήκαν απλώς στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν και πολλοί από αυτούς καταδικάστηκαν σε θάνατο. Είδαμε μαζικές ποινές να επιβάλλονται, δημοσιογράφοι να συλλαμβάνονται όπως όλοι γνωρίζουμε και ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού ε, πεινάει, ε, δεν έχουν πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα όταν αυτή απαιτείται. Είναι απαράδεκτο αυτό. Πρέπει να είμαστε πολύ σκληροί εναντί της Αιγύπτου Πρέπει να βοηθήσουμε τις Αιγυπτιακές αρχές, αλλά μόνο αν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και μόνο αν σταματήσουν αυτές τις εκτελέσεις και την επιβολή θανατικών ποινών και αν απελευθερώσουν πολιτικού κρατούμενους. Αν η Αίγυπτος είναι σημαντική εταίρο για μα, όλοι το λένε αυτό άλλωστε εδώ στην Ολομέλεια, τότε για αυτή την περιπτώση θα πρέπει η Αίγυπτος ε, να φροντίζει και για τα ανθρώπινα όντα που υποφέρουν και χρειάζονται τη βοήθειά μα. Πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη αδιάσταση του του προβλήματος Αιγύπτου. Δίνω το λόγο για την τελική παρέμβαση, την είπατε εκπρόσωπο, την Αντιπρόεδρο, την κυρία Μογκερίνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους σας ε, τα μέγιστα για τη συζήτηση αυτή και για την αξιολόγηση της παρουσίασης, ε, της παρουσίας, της παρουσίας μου εδώ στην Ολομέλεια. Πρέπει πραγματικά να αναθερήσουμε τις διαδικασίες της Ολομέλειας. Όχι για μένα, αλλά για σας τους Ευρωβουλευτές. Για μένα, για μένα δεν είναι μόνο καθήκον. Δεν ξέρω σε τι έχετε συνηθίσει, αλλά όταν υπάρχει μια συζήτηση που αφορά δικές μου αρμοδιότητες είναι καθήκον μου να παρίσταμαι. Επίσης είναι πολύ ενδιαφέρουσα και είναι πραγματικά θελκτικό να παρακολουθεί κανείς τη συζήτηση. Είναι πολύ γόνιμο και επικοδομητικό και επιτρέψτε μου επίσης να προσθέσω ότι θα είμαι παρούσα και εδώ αύριο το πρωί και θα είμαι μαζί σας και σε σχέση με την ακρόαση, όταν είπα ότι θα συνεργαστώ με το Ευρωκοινοβούλιο, το εννοούσα και είναι πραγματικότητα αυτό. Δεν χρειάζεται να με εγκομιάζετε γι' αυτό. Είναι κανονική διαδικασία, κανονική κατάσταση των πραγμάτων και καθήκων μου. Πρέπει να βρούμε ένα πιο ορθολογικό τρόπο για τη διεξαγωγή του κοινοβουλευτικού έργου και τη διεξαγωγή των ολομελιών όμω. Και τούτου λεχθέντος πιστεύω ότι η συζήτηση για αυτό το θέμα καταδεικνύει ότι είναι το μόνο από τα τρία ψηφίσματα που είχατε εφέτος, που υπήρξαν εφέτος, που δίνει μια τέτοια προοπτική, μια αξιολόγηση, αποτίμηση μεταξύ δύο διαφορετικών θεμάτων. Πρώτον, του περιφερειακού ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει και έχει διαδραματίσει η Αίγυπτος σε σχέση με την μεσανατολική διεργασία και διαδικασία και πολλά από τα θέματα που έχουν κέρια σημασία για μας μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Από την άλλη πλευρά η εσωτερική μεταβατική περίοδος που ε, περνά αυτή τη, στιγμή η Αίγυπτος πρέπει να ε, υποστηριχθεί για τις ε, κατευθύνσεις που αναφέρθηκαν από εσά για τις, τον σεβασμό των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η ίδια η Αίγυπτος και είναι μια μεταβατική περίοδος κατά τα άλλα αυτή. Δεν θα συμφωνούσα με εκείνους που λένε ότι η αραβική άνοιξη περνά σε ένα αραβικό χειμώνα. Πρώτον, δεν θα ήταν σωστή αυτή η περιγραφή για την Αίγυπτο με την έννοια, με την περιγραφή αραβικού χειμώνα. Δεν είναι λοιπόν Ισλαμικός χειμώνας. Και επίσης όταν έχουμε προσέγγιση αυτών των χωρών πολλές φορές ε, δεν είμαστε πάρα πολύ γενναιόδοροι. Πολλές φορές πήρε δεκαετίες ε, για ευρωπαϊκές χώρες να ολοκληρώσουν μεταβατικές ε, περιόδους εκδημοκρατισμού τους και αυτό δεν πρέπει να είναι κάτι ξεχωριστό και αντιφατικό για την Αίγυπτο. Και βλέποντας το ιστορικά Υπάρχει αυτή η προοπτική. Μπορεί να είναι δυσχερές το εγχείρημα, αλλά δεν θα έπρεπε να, έπρεπε να πούμε ότι κλείνει κάθε προοπτική με αυτή την ε, ε, κατάσταση. Και γι' αυτό βρισκόμαστε ακόμα στην Αραβική Άνοιξη. Και πολλές φορές υπάρχουν πτυχές ε, που μπορεί να θεωρηθούν επιτυχής για, την, για μια μεταβατική τέτοια περίοδο. Και σε πολλές περιπτώσεις ε, όταν βλέπουμε την ανάδυση μιας κοινωνίας πολιτών που αναδύεται αυτό είναι πραγματικό και αξία για μια τέτοια χώρα. Πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω μια πιο ας το πω έτσι εμβαθυμένη ενδελεχής ανάγνωση των τεκτενομένων σε αυτή τη χώρα. Και επίσης ε, πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη ότι έχουμε επεκταθεί επαρκώς όμως ε, θα ήθελα να αναφέρω δύο επιπλέον πράγματα. Αφενός υπήρξε μια συγκεκριμένη περίπτωση που αναφέρθηκε από πλευράς Ευρωβουλευτών και θέλω να το αναφέρω αυτό διότι συζήτησα αυτή την περίπτωση προχθές στο Δουβλίνο την περίπτωση του Ιμπραχήμ Αλάουα και ενός ε, Ιρλανδού πολίτη που βρίσκεται στην ε, Αίγυπτο ε, υποκράτηση παρακολουθούμε με τα τελευταία στοιχεία το τι συμβαίνει με τον άνθρωπο αυτό και με τις υπηρεσίες μας και με τις Ιρλανδικές αρχές και τους αρμοδίους. Αυτά σε σχέση με το αν αναφέρω ένα θέμα ή ένα άλλο θέμα αυτό σε σχέση με τις αρχές της Αιγύπτου, με τα στοιχεία τα οποία υποβάλλονται, ακόμα δεν είχα μια επίσημη συνάντηση με τις αραβικές αρχές, με ε, την αραβική κυβέρνηση. Είχα κάποιες επαφές υπό διαφορετική ιδιότητα, αλλά όχι υπό το σημερινό μου αξίωμα ως υπά του εκπροσώπου. Και έτσι λοιπόν έχουμε και μηνύματα τα οποία πρέπει να, να ληφθούν υπόψη δεόντως. Πράγματι θα σχεδιάσω και θα προγραμματίσω μια τέτοια συνάντηση ώστε να δούμε τι μπορεί να γίνει σε σχέση με τις ε, αρχές της Αιγύπτου. Ακολουθώντας τις ε, προτάσεις ε, της μεγάλης πλειοψηφίας των Ευρωβουλευτών πρέπει να βρούμε μια σωστή ισορροπία εμπλοκής μας σε άμεσο επίπεδο, σε ένα επίπεδο διαλόγου με τις Αιγυπτιακές αρχές για να ευδοκιμήσουν αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Έχω λάβει 7 προτάσεις ψηφίσματος που θα ψηφιστούν αύριο, 5η. 15 Ιανουαρίου στις 12.30. Πριν από την επόμενη και τελευταία συζήτηση θέλω να σας ευχαριστήσω την Πρόεδρε μου για τη σημερινή σας δουλειά και για την ε,